Είχαμε την τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Λίμπε τη Δευτέρα και την Τρίτη και τώρα την Πέμπτη, αμέσως μετά την Ολομέλεια. Οπότε ας ξεκινήσουμε μια ώρα αρχίτερα και να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Καταρχήν να σας θυμίσω ότι έχουμε ψηφοφορία απόψε. Οπότε θα πρέπει να έχετε όλες σας τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Όποιος έχει ξεχάσει την ηλεκτρονική του κάρτα στην αίθουσα της Ολομέλειας, να καλέσει τον βοηθό του να τρέξει γρήγορα να τη φέρει. Then we move to point number one. Περνάμε στο σημείο 1. Ε, έγκριση της μερίσης διάταξης. Έχουμε μια πρόταση του εισηγητή για το σημείο 6, δικαίωμα ενημέρωση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Η εισηγήτρια είναι η Συνάδελφο Σίπελ. Αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση της ε, συνεδρίασης ΛΥΜΠΕ. Μετά το σημείο 7, η απουσία Διαβίβαση από το Συμβούλιο των Σχετικών Εγγράφων που αφορούν την πρόσβαση, την προσχώρηση μάλλον της Βουλγαρία και τη Ρουμανία στο σύστημα Σέγγεν, σήμερα θα κάνουμε μόνο μία δεύτερη ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θέμα. Το σχέδιο έκθεση θα υποβληθεί μόλι θα έχουμε στη διάθεσή μα τι πληροφορίε. επιμένουμε γι' αυτό. Έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο με το Συμβούλιο για να του θυμίσουμε τη σημασία του να έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα αυτά, γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ο εισηγητής θα μας ενημερώσει για το πού βρίσκεται η κατάσταση, ο κ. Κουέριο, και μετά έχουμε την πρόταση για οδηγία για την ε, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, την παιδική πορνογραφία. Είναι ε, απόφαση πλαίσιο. του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων που έχει αναβληθεί για τη συνεδρίαση για τις 14 Φεβρουαρίου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται με λύση διάταξη. Τώρα, η πλειοψηφία των συντονιστών συμφώνησε να αναβάλει τη συνεδρία των συντονιστών που είχε προγραμματιστεί για σήμερα. Ναι. Και για τα επίγοντα θέματα θα ακολουθηθεί η γραπτή διαδικασία. Θα ξεκινήσει αμέσως. Οπότε, περνάμε στα πρακτικά της περασμένης συνεδρίασης. Δεν έχετε παρατηρήσεις? Όχι. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Ας πάμε στο σημείο 4 που αφορά την διαδικασία νέας αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας. Εδώ έχουμε εισηγήτρια τη συνάδελφο Βερονίκ Ματιέ. Θα πρέπει να έχετε υπόψη για το θέμα αυτό που αποκαλείται ενιαία άδεια. Στην τελευταία μας συνεδρίαση αποφασίσαμε να περιορίσουμε την ψηφοφορία μας στο τμήμα του νομοθετικού κειμένου που καθορίζει την απόρριψη από την Ολομέλεια της πρότασης για ενιαία άδεια που μας έστειλε η Κομισιόν. Οπότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Επιτροπή Απασχόλησης, Απασχόλησης ή Εμπλόη που είναι συνδεδεμένη με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 50 του κανονισμού του Κοινοβουλίου, αμφισβήτησε την ερμηνεία της ΛΥΜΠΕ για το άρθρο 56, το οποίο είχε γίνει αντικείμενο συζήτηση στη Δευτέρα το απόγευμα. Οπότε, η Επιτροπή Απασχόλησης, μέσω του Πρόεδρου της, υπέβαλε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριο Μπούζεκ, ένα αίτημα για μια διευκρινιστική τελική ερμηνεία από το αρμόδιο σώμα. Αυτό δηλαδή που ερμηνεύει τους κανόνες, τον κανονισμό του Κοινοβουλίου που είναι η, εκθέση, η Επιτροπή ΑΦΚΟ. Άρθρο 56, παράγραφος 3. Αφού αναμένουμε λοιπόν την συνέχεια που θα δοθεί σε αυτό το αίτημα, σύμφωνα με τον κανονισμό πάντα, θα πρέπει να υποβάλουμε την έκθεσή μας στην Ολομέλεια πριν από το τέλος δίμηνη προθεσμίας που προέβλεπε το ίδιο άρθρο. Οπότε προτείνω να προχωρήσουμε με την ψηφοφορία όπως έχουμε συμφωνήσει για το άρθρο 7 και 16.1 της πρότασης της Επιτροπής, όπως είχαμε συμφωνήσει στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Βλέπω ένα διαδικαστικό. Ο κύριος Μωράης, ναι, όχι, όχι. Ο κύριος Μωράης. Πρόεδρε, για την τελευταία σας παρατήρηση για την ψηφοφορία. Θα ήθελα να ζητήσω την κατανόηση της Επιτροπής σας για το θέμα της νομικής συμβουλής από την ΑΦΚΟ εγώ κατάλαβα πως αυτή θα είναι διαθέσιμη την επόμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει ακόμα η γνωμοδότηση. Για να είμαστε συνεπείς λοιπόν σε αυτό που ζητήσαμε, γνωρίζουμε πως ίσως η Επιτροπή να δεσμευτεί από αυτή τη νομική συμβουλή ή όχι όταν θα μας έρθει την επόμενη εβδομάδα και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να είμαστε συνεπείς και να ζητήσουμε για μια απλή ψηφοφορία, να μην αρχίσουμε συζήτηση επί της διαδικασίας, δεν το επιθυμούμε αυτό. Θέλουμε όμως μια ε, απλή ψηφοφορία πριν μπούμε στις ψηφοφορίες επί της ουσίας για το θέμα της αναβολής μέχρι ότου να έχουμε στα χέρια μας την νομική γνωμοδότηση. Και πάλι δεν θέλω να ξεκινήσω ε, διαδικαστική συζήτηση, απλώς θα ήθελα να ψηφίσουμε για το κατά πόσο θα πρέπει ή όχι να αναβάλουμε βάλουμε την ψηφοφορία επί της εκθέσεως μέχρι ότου να έχουμε την νομική γνωμοδότηση. Και δεν θα ήθελα να καθυστερήσουμε, να προχωρήσουμε άνευ συζητήσεως. Και μετά αναλόγως του αποτελέσματο να προχωρήσουμε. We have heard a proposal by the S&D Ακούσαμε μια πρόταση από τον συντονιστή των σοσιαλιστών, τον κύριο Μωράης, ο οποίος προτείνει χωρίς καθυστέρηση να ψηφίσουμε για αυτό το διαδικαστικό θέμα που είναι μια πρόταση για αναβολή της ψηφοφορίας. Κύριε Ταβάρη, θέλετε να κάνετε διαδικαστικό. Ωραία, λοιπόν, τότε ψηφίζουμε επί της πρότασης για αναβολή της ψηφοφορίας εν αναμονή της νομικής γνωμοδότησης που ζήτησε η Επιτροπή Απασχόλησης. Μέσω αυτής της διαδικασίας που σας εξήγησα, την επιστολή του κ. Μπούζεκ, ο οποίος παρέπευσε το θέμα στην Συνταγματική Επιτροπή, για μια διευκρινιστική ερμηνεία όσον αφορά το άρθρο 56. Θα ψηφίσουμε λοιπόν για την πρόταση. Αναβολή λοιπόν της ψηφοφορίας μέχρι ότου να έχουμε την νομική γνωμοδότηση. Αυτή την πρόταση ψηφίζουμε τώρα, εντάξει. Ψηφίζουμε. You got problems? Eh, now you, you, will be telling who, who... Έχετε πρόβλημα να μου πείτε αν κάποια νόη κάρτα δεν δουλεύει ή λείπει. Τέλος της ψηφοφορίας. 19 συν 30 πλην. Ένας πρέπει να μετρηθεί στους συν 20-30 λοιπόν, οπότε θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία όπως είχαμε συμφωνήσει. Στις τροπολογίες δηλαδή, κανονικά. Σύμφωνοι. Άρθρο 7, παράγραφος 1. Ψηφίζουμε. Now the vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. 45 plus, be against. It's a... 45 υπέρ, 3 κατά, εγκρίνεται. Άρθρο 16, παράγραφος 1. Ψηφίζουμε. Apparently there is one plus PP. There is... Ένας παραπανήσιος από το ΕΛΚ ψηφίζει. So, we got... The vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. Yes. It's 46 plus. 46 υπέρ, 2 κατά. Άντε 47 υπέρ. Γιατί ο κύριο Κάσμαν δεν μπορεί να ψηφίσει με την εικονική του κάρτα. Άρα είναι 47. Ε, υπέρ εγκρίνεται. I remind you that the new deadline... Να θυμίσω ότι η νέα προθεσμία... Yes, I see. Moving to point number five. Διακοψε ο Πρόεδρος. Περνάμε στο σημείο 5. Eurodac για τη σύγκριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων αναδιατύπωση. θα κάνουμε μια ψηφοφορία προς ανατολισμό για τη δημιουργία του συστήματος Eurodac, για το οποίο είναι υπεύθυνη η συγγήτρια, η κυρία Μακοβέη. Εμείς, θα θυμάστε, δώσαμε εντολή στην εισηγήτρια για τη συζητήση με το Συμβούλιο. No, I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 Θα ψηφίσουμε δυνατά σα τη χειρό. Έχετε του ε, κατάλογου ψηφοφορία. Ωραία, ευχαριστώ. Amendment 29. Those in... Τροπολογία 29, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 34 δεν την ψηφίζουμε, 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 37 και 38 είναι ταυτόσιμες. Τες ψηφίζουμε από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ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 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα ψηφίζουμε για τα εκτιμώντας και τις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έτσι καταπίπτει η τροπολογία 25 και πάμε στη συμβιβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 καταπίπτει. Συμβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 καταπίπτει. Και τώρα ψηφίζουμε για τις παραγράφους του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος. Οι τροπολογίες 20 και 21 και 22 είναι ταυτόσημα στη ψηφίζουμε από κοινού. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογίες 23 και 24 έχουν αποσυρθεί. Οπότε ψηφίζουμε για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ. Καλύτερα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για τα πρακτικά ψηφίζουμε. Τέλος πληροφορίας. Ένας παραπανήσιος πάλι στο ΕΛΚ. Τέλος της πληροφορίας. It's 44 favor, against. υπέρ, 3 κατά. 3 αποχές, οπότε εγκρίνεται. Έχουμε την ψηφοφορία προς ανατολισμό μας, κυρία Μακοβάη. Ευχαριστούμε. Το έξι έχει ε, αναβληθεί και τώρα περνάμε στο 7. Το 7 που αφορά την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σέγγεν στις δημοκρατίες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Ακούσουμε πού βρίσκεται η κατάσταση, ποια είναι η κατάσταση πρόοδου Παρακαλώ, ησυχάστε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Make it shorter for all of us. Και να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. I think we, we should be concerned about our way home <laughs> Thursday evening. So... Για να πορευτούμε και για τα σπίτια μας. Πέμπτη απόγευμα είναι, λέει ο πρόεδρος. Κύριε Κοέλιο, παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ας ακούσουμε τον κύριο Κουέλιο, τον εισηγητή μας. Thank you so much, President. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακάλεσα τις υπηρεσίες να διανύμουν σε όλα τα μέλη ένα σύντομο έγγραφο που περιγράφει την κατάσταση όσο έχει τώρα. Ελπίζω δε ότι διανέμεται αυτή τη στιγμή. Πάντως, είναι μια μοναδική κατάσταση. Εδώ τονίζω τρία πράγματα. Πρώτα σχετικά με την ταχεία διαδικασία. Ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους που συμφώνησαν να εφαρμοστεί κατ' εξαίρεση αυτή η ταχεία διαδικασία. Δηλαδή, χρήση μόνο του εγγράφου στα αγγλικά για να αποφευθούν καθυστερήσεις λόγω μεταφράσεων ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να εκδώσει γνωμοδότηση πριν από το Συμβούλιο Τζάι, Δικαιοσύνη και Εσωτερικών, για τις 20, που προβλέπεται στι 24 και στι 25. Πάντως, όπω ξέρετε όλοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει λάβει τα έγγραφα που ζήτησε. Και εννοώ τις εκθέσεις εξελίξεως για τη Βουλγαρία και την Ρουμανία, καθώς και τις συστάσεις που έχουν γίνει για τις χώρες αυτές και τις προφορίες για το λεγόμενο state of play, σχετικά δηλαδή με το πού βρίσκονται οι χώρες αυτές με την εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Ξέρουμε επίσης ότι το Συμβούλιο Δικαιοσύνης των Τελικών του Φεβρουαρίου δεν σχεδιάζει να λάβει αποφάσεις για την, για, τις, ε, για την προσχώρηση στο σύστημα Σέγγεν των δύο χωρών. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος για να διατηρηθεί η ταχεία διαδικασία. Προτείνω λοιπόν να ακολουθηθεί η συνήθις διαδικασία με ε, μετάφραση του κειμένου σε όλες τις γλώσσες εργασίας. Δεύτερο, πρόσβαση στα έγγραφα. Η συνθήκη προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να μπορέσει να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο του στην διαδικασία αυτή. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου λένε τα ίδια πράγματα. Εσείς κύριε Πρόεδρε, με επιστολή σας της 16ης 12 του προηγουμένου έτους ζητήσατε από το Συμβούλιο να διαβιβάσει τις σχετικές εκθέσεις. απάντηση λάβαμε πλέον των 40 ημερών αργότερα και η οποία απάντηση έλεγε ότι τα έγγραφα που είχαν ζητηθεί μπορούσαν να τεθούν υπόψη του Προέδρου, των συντονιστών και του εισηγητού. Και αυτό σε ασφαλές γραφείο στα κτίρια του Συμβουλίου. Η επιστολή αυτή τονίζει επίσης ότι δεν θα πρέπει να γίνει άμεση αναφορά στο περιεχόμενο των εγγράφων αυτών σε οποιαδήποτε συνεδρίαση. Που μας αφήνει με ένα πρόβλημα. Δηλαδή, τι θα γράψουμε εν τέλει στην έκθεση για τις δύο αυτές χώρες, εάν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε πληροφορία που θα έχουμε ε, λάβει από τις εκθέσεις αυτές. Εδώ επιθυμώ να τονίσω και πάλι ότι το Συμβουλίο προσφέρει λιγότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα από ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια το 2007 όταν το Κοινοβούλιο είχε γνωμοδοτήσει για εννέα τότε χώρες Τσεχία, ε, Λιθουανία, τις άλλες βαλτικές χώρες και ούτω καθεξής. Δεν έχει λοιπόν κανένα νόημα απολύτως τώρα, διότι τώρα το Συμβούλιο Υπουργών διαβιβάζει λιγότερες πληροφορίες από αυτές που μας διαβίβαζε προτετραετίας πριν από τη συνθήκη της Αβώνας δηλαδή. Το τονίζω αυτό, διότι θεωρώ το γεγονός αυτό απαράδεκτο. Το Συμβούλιο μας φέρεται κατά χείριστο τρόπο, χειρότερο από ό,τι έκαναν πριν από την ε, θέση σε ισχύ της συνθήκης της Αβώνας. Και τώρα που έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνα, το Κοινοβούλιο έχει περισσότερα δικαιώματα και πρέπει αυτά να γίνονται σεβαστά. Το 2007 και μάλιστα τα έχω γραπτός αυτά και τα έχω γράψει και στο έγγραφο που σας έχω διανύμει, το Συμβούλιο επέτρεψε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών να εξετάσουν τις εκθέσεις προόδου, τις πλήρες εκθέσεις προόδου για τις υποψήφιες εκείνες χώρες και εκ παραλίλου, εκ και δεν ήταν άλλη επιλογή αυτή και τα συμπεράσματα σχετικά με τις εξελίξεις εκείνες που αποχαρακτηρίστηκαν τα συμπεράσματα αυτά, τα πορίσματα αυτά και διαβιβάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, τελευταίο σχόλιο. Νομίζω, ελπίζω, ότι θα προσφέρει τελικά πρόσβαση στα έγγραφα το Συμβούλιο. Στην συνάντησή μου όμως με τους σκιώδης τέθηκε μια ερώτηση. Εάν το Συμβούλιο δεν διαβιβάσει τις εκθέσεις, για παράδειγμα μέσα στο 2011, θα περιμένουμε για πάντα οι σκιώδεις ηγητέ συμφώνησαν μαζί μου ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε για πάντα. Άρα θα πρέπει να αποφασίσουμε, θα πρέπει να εγκρίνουμε μία ε, προθεσμία, μία ημερομηνία, μέχρι την οποία θα περιμένουμε να μας διαβαστούν οι εκθέσεις από το Συμβούλιο. Εάν όμως δεν λάβουμε τίποτε και εκπνεύσει αυτή η προθεσμία, θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε εάν δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τις συνθήκες ασφάλειας. Δηλαδή θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε ε, γνωμοδότηση. Με αυτή τη γνωμοδότηση όμως ολοκληρώνει τη διαδικασία του Κοινοβουλίου και δεν δίνει την ευκαιρία στο Συμβούλιο να πει ότι δεν μπορεί να λάβει απόφαση διότι αναμένει τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό προτείνω την ε, προθεσμία, προθεσμία της Δευτέρας Μαΐου και ελπίζω, ελπίζω κύριε Πρόεδρε να μας στείλει τα έγγραφα για τη Ρουμανία και Βουλγαρία πριν από την ημερομηνία αυτή ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την διαδικασία γνωμοδοτήσεως. Αν όμως δεν συμβεί αυτό, να μην περιμένουμε περαιτέρω περισσότερο από τις 2 Μαΐου και να προχωρήσουμε όπως σας είπα και όπως είπα στην ε, πρότασή μου αυτή συμφωνούν και οι σκιώδεις Ευχαριστώ για την διαυγή εξήγηση της ε, κατάστασης όπως ε, διαγράφεται αυτή τη στιγμή. Σας υποστηρίζει νομίζω όλη η Επιτροπή και η Γραμματεία και ο Πρόεδρος σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ακούσουμε ορισμένους βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο. Πρώτος κύριος Ένσιο. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το εξαίρετο το έργο για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το διέξοδο όπου μας έχει οδηγήσει το Συμβουλίο. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι φυσιολογικό να βρισκόμαστε σε τέτοια κατάσταση. Εξ ονόματο ε, της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να πω ότι είμαστε 100% ε, υπέρ τη στρατηγική που προτείνεται κύριε Κοέλιο. Ίσως ε, εγώ να είμαι και κάποιος ε, κάπως ε, έτσι επαναστάτη στη σκέψη μου. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά όχι να αφήνουμε το Συμβουλίο να κάνει ό,τι του κατεβαίνει. Και με την ησυχία του είναι καλό να βρούμε με έναν νομική όδο, ώστε η συνθήκη της Λισαβόνας και οι νέε αρμοδιότητε του, ε, του Κοινοβουλίου με να γίνονται σεβαστέ από το Συμβούλιο. Εγώ συνομίλησα με τον εισηγητή και μου είπε πω δεν ήταν δυνατόν να φέρουμε το, το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά ίσω θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε τη γνώμη του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το ζήτημα αυτό. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να αφήσουμε το Συμβούλιο να κάνει ό,τι θέλει, γιατί πραγματικά είναι σαν να δεχόμαστε ένα χαστού και εμείς και η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρινέσκου. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω εσάς κύριε Σιγητά, να ευχαριστήσω τους ε, συντονιστές, τους και συζητητές, αλλά και όλα τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που δέχτηκαν να αλλάξουν την διαδικασία. Δέχτηκαν την ε, ταχεία διαδικασία ώστε να μπορέσουμε να εκφράσουμε την ψήφο μας πριν την ε, το Συμβούλιο Τζάι στις 24 Φεβρουαρίου. Δυστυχώ αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε και αυτό λόγω τη τάση που, που κρατά το Συμβούλιο. Στην ομάδα επαφή την τελευταία εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα υιοθετήθηκε η τεχνική έκθεση για τη Ρουμανία, δηλαδή ω το τεχνικό επίπεδο η Ρουμανία έχει ήδη πληρώσει όλα τα κριτήρια. Κύριε Πρόεδρε, απαιτήσατε τα έγγραφα από πλευρά Συμβουλίου ε, και η Ρουμανία και η Βουλγαρία ζήτησαν να δημοσιευθούν αυτά τα έγγραφα ώστε να μπορέσουν να σταλούν και στο Κοινοβούλιο, αλλά δυστυχώ το Συμβούλιο αρνείται. και με τη στάση του αυτή δεν κάνει παρά να καθυστερεί τη λήψη μιας απόφασης. Γιατί αυτό το αίτημα από διαβάθμιση των εγγράφων αυτών υπάρχει στην ημερήσια διάταξη της Κορεπέρ μόνο από τις 9 Φεβρουαρίου. Για τις 9 μάλλον Φεβρουαρίου. Η Ρουμανία λοιπόν ε, σκέφτεται να στείλει όλες τις επίσημες εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί δεν μπορούμε να σε περιμένουμε παόριστο όπως έλεγε και ο εισηγητής στην παρέμβασή του. Δεν μπορούμε να περιμένουμε παόριστο τη θέση του Συμβουλίου που θα μπορούσε να φτάσει πολύ καθυστερημένα και άρα προσπαθούμε να διερευνήσουμε κάθε δυνατότητα για να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες στο Ευρωκοινοβούλιο, ούτω ώστε τα μέλη της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ και του Ευρωκοινοβουλίου να μπορέσουν να ψηφίσουν έχοντας εν γνώση μάλλον της υπόθεσης. Και ένα τελευταίο αίτημα, αυτό η προθεσμία της Δευτέρας Μαΐου, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ μακρινή προθεσμία. Εγώ θα ήθελα να, να θεωρηθεί αυτή η ημερομηνία. Αν για παράδειγμα το Συμβούλιο δεν μας στείλει τα έγγραφα αυτά, και σε περίπτωση όπου η Βουλγαρία λάβει θετική ψήφο στις εκθέσεις της, νομίζω πως το αργότερο το Μάρτιο μπορεί το Κοινοβούλιο να βρει τρόπο για να ψηφίσει την ε, έκθεση αυτή. Τώρα, σε αυτές τις εκθέσεις μέσα περιλαμβάνεται και η επιστολή των δύο υπουργών. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Πώς ένα έγγραφο το οποίο είναι δημόσιο και έχει δημοσιευθεί στα πρωτοσέλιδα έχει διαβαθμιστεί σε αυτή, στην αίθουσα των ε, διαβαθμισμένων εγγράφων. Εγώ όταν άνοιξα το φάκελο βρήκα και αυτές τις επιστολές. Διαρωτώμε σε τι χρησιμεύουν όλες αυτές οι επιστολές. Φαντάζομαι πως όλοι οι βουλευτές γνωρίζουν τις επιστολές αυτές. Για, τι λοιπόν συμβαίνει αυτό. Είναι κάτι μυστήριο. Θα ήθελα να βρούμε τη λύση στο ένιγμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο Σκιώδης από την άλλη θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Κάρλος Κοέλιο για όλες τις προσπάθειες που έχει καταβάλει και πραγματικά ήταν εξαιρετική δουλειά που έκανε και τα έγγραφα που έχει προετοιμάσει είναι πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι έχει δώσει όσο μεγαλύτερη ευελιξία μπορούσε στη συζήτηση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Άρα, ως και ό,τι ναι, χαίρομαι και είμαι πολύ ικανοποιημένη με τη γραμμή που προτείνει. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση στο σημείο αυτό σε δύο επίπεδα συζήτηση. Καταρχά. το τι θα κάνουμε με το συγκεκριμένο φάκελο, με τη Ρουμανία και την ε, πρόσβαση, την ε, προσχώρηση του Σέγγεν. Δεν θα λάβει ε, απόφαση το Συμβούλιο, από ό,τι φαίνεται, και νομίζω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε τη Δευτέρα Μαΐου ως προθεσμία, γιατί μπορούμε να ψηφίσουμε πριν ε, την Δευτέρα Μαΐου, άρα μπορεί να λάβει το Συμβούλιο την απόφαση να λάβει την απόφαση να δεχτεί τις χώρες αυτές. Άρα εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Κατά δεύτερον, έχουμε και το θέμα επί της αρχής, σε ό,τι αφορά τη θεσμική συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Πριν από δύο εβδομάδες, ούτε καν δύο εβδομάδες, δέκα μέρες, ήμουν με τους συντονιστές και την ηγεσία της Άλντε στη Βουδαπέστη. Συναντηθήκαμε με τον Βίκτορ Όρμπαν, τον Πρωθυπουργό, τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και θέσαμε το ζήτημα αυτό τότε μας διαβεβαίωσε, μας είπε ότι κατανοεί απόλυτα ως ε, βουλευτής, ε, ως πρώην βουλευτής της χώρας τους, ότι φυσικά οι βουλευτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα πρωτού ψηφίσουν. Αυτό είναι φυσιολογικό, μας είπε. Ωστόσο, η ουγγρική αντιπροσωπεία και η απάντηση που μας έδωσε τελικά ήταν κάθε άλλο παρά ικανοποιητική. Ο κ. Ντόουλα έστειλε μια επιστολή προς τον κ. Ορμπάν μια και βιαζόμαστε όμως πλέον, θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη αυτή με το Συμβούλιο, γιατί όντω φαίνεται ότι το Συμβούλιο θέλει να θέσει ένα προηγούμενο, να δημιουργήσει προηγούμενο. Και τι το Κοινοβούλιο μπορεί να έχει συναπόφαση, να έχει και δικαίωμα ψήφου, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι εξίσου σημαντικό όσο και το Συμβούλιο και παραμερίζεται, βραγκονίζεται και δεν νομίζετε. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο, γιατί υπάρχει και η θεσμική διάσταση του θέματος. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από τον πρόεδρο Μπούζεκ προσωπικά ή μέσω επιστολή να έρθει σε επαφή με το Συμβούλιο και να το διαλευκάνει το θέμα. Και μάλιστα με τρόπο δίκαιο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστώ κυρία Βέμπερ. Αυτός ε, αυτό ακριβώς αποφάσισαν και οι συντονιστές. Και βλέπω τώρα ότι ο κατάλογος των ε, βουλευτών που θέλουν να πάρουν το λόγο μεγαλώνει. Δεν βλέπω όμως να υπάρχει οποιαδήποτε διαφωνία. Όλοι οι συνάδελφοι επιμένουν στα θέματα που αναφέραμε, επιμένουν στο θέμα του σεβασμού που πρέπει να δείχνει το Συμβούλιο προς το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των καθηκόντων του Κοινοβουλίου. Άρα θα σας παρακαλούσω να μας βοηθήσετε να μην ε, μακρηγορούμε ιδιαίτερα. Η κυρία Ιντφέλτ έχει το λόγο. Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Συμφωνώ με όλα όσα ακούστηκαν ως τώρα. Όλα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι και καλωσορίζω τη γραμμή που επέλεξε ο εισήγητης. Να προσθέσω όμως ότι δεν είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκείνο που έχει δικαίωμα να γνωρίζει, να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Όχι, οι λαοί της Ευρώπης, ο λαός της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας. Και μου προκαλεί αποτροπιασμό το γεγονός ότι βλέπω ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν θέσει το θέμα της προσχώρησης στο Σέγγεν ως θέμα εσωτερική πολιτική Είναι πραγματικά ιδιαστικό αυτό και νομίζω ότι δημιουργεί προηγούμενο. Δεν νομίζω ότι η συζήτηση αυτή θα πρέπει να βρωμίζεται με ε, επιχειρήματα που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με το Σέγγεν. Οι εθνικέ κυβερνήσει να αναλαμβάνουν τι ευθύνε του. Και γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζω την πρότασή σα να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία θα ακολουθεί τα σωστά κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται ισότιμα προ όλε τι χώρε και για όλου του πολίτε. Η επόμενη ομιλήτρια, η ε, κυρία Νελτσέβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή τον κύριο Κοέλιο και να συμφωνήσω μαζί του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. на досието за Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή και για το γεγονός ότι έθεσε σαφώς τις σχέσεις με το Συμβούλιο και ε, μας εξήγησε και πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Και θα ήθελα να προτείνω να ακολουθήσουμε τη στρατηγική που προτείνει, να θέσουμε δηλαδή μία ημερομηνία, καταλεκτική. Είναι απαραίτητο αυτό. Πρωτού γνωμοδοτήσουμε βάση των εγγράφων και των ε, πληροφοριών που θα έχουμε λάβει. Ιδάλλως, όλα τα υπόλοιπα είναι εικασίες. Και θα γίνουν τέτοιες εικασίες και στην ε, Βουλγαρία και στην Ρουμανία. Αυτό προκαλεί ασφαλώ σύγχυση. Και είναι πραγματικά περίεργο το γεγονός ότι δεν έχουμε τελικά ακριβείς πληροφορίες στην διάθεσή μας. Αυτές οι σχέσεις λοιπόν μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου είναι ιδιαίτερα σημαντικές και πρωταρχικό θέμα είναι η θεσμική συνεργασία. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν πιο πολλές πληροφορίες για το πώς έχουν τα πράγματα Θα πρέπει να λεφθούν υπόψη οι αρμοδιότητε που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επόμενο ομιλητέ, ευχαριστώ. Ω συντονιστή του ΕΛΚ, θα ήθελα να τονίσω ότι το ΕΛΚ υποστηρίζει την προσχώρηση τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία στην ζώνη Σέγγεν και ο κύριο ο κύριος ε, Κοέλιο εξέφρασε την ε, άποψη και την τοποθέτηση όλη τη ομάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ και θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι εξίσου σύντομη. Συμφωνώ με την κυρία Βέμπερ ότι το θέμα αυτό είναι... έχει δύο πλευρές. Καταρχάς το θέμα της ουσίας. Δεν θέλω να αναφερθώ θέμα θέματα ουσίας γιατί πολλά ακούσαμε ήδη ως προς αυτή τη διάσταση. Έχω την εντύπωση η κατάσταση είναι η παρόμοια με την κατάσταση του 2007, με την τελευταία φορά που προσχώρησαν τα νέα κράτη-μέλη στην ζώνη Σέγγεν. Αυτό που είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό είναι ότι υπάρχει τέτοια παρακράτηση πληροφοριών ακόμα και μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Άρα θεωρώ ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένο, Πρόεδρε, να ζητήσετε διευκρινήσεις, γιατί η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα έρθει αντιμέτωπη με την ίδια κατάσταση πολλές φορές. Αλλά θεωρώ ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένο να αναλάβει τέτοια δράση και ο Πρόεδρος Μπούζεκ. Άρα να ζητήσω από τους συντονιστές να αποφασίσουν ποιος θα ζητήσει τις διευκρινήσεις στην τρέχουσα κατάσταση. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι η τελευταία φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση και είναι πολύ σοβαρό το θέμα και θα πρέπει εξ αρχής να λυθεί σωστά. Να διευκρινιστεί τι γίνεται με τις πληροφορίες που δίνει το Συμβούλιο. Και δεν είναι θέμα Προεδρίας, είναι θέμα Συμβουλίου. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, έχετε δίκιο και το έχουμε συζητήσει αυτό στους συντονιστές και επιμένουμε στο θέμα αυτό. Ζητήθηκε από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Μπούζεκ, να ε, θέσει το θέμα αυτό στο Συμβούλιο εξ ονόματος του συνόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Ταβάρες. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και εγώ, γιατί είμαι σκιώδης, εισηγητής, αλλά Μιλώ εξ ονόματος της πολιτικής ομάδας μου ως συντονιστής και θα ήθελε και ο κ. να αναφέρει ότι και τα δύο θέματα τα οποία διακυβεύονται εδώ το γεγονό ότι δίνεται πολιτικό χαρακτήρα στην προσχώρηση του, στη ζώνη Σέγγεν τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και οι, οι υπόλοιπε δυσκολίε που προκύπτουν για το δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου λόγω παρακράτησης των ε, εγγράφων αυτών είναι θέματα τα οποία μας δυσαρεστούν και θα θέλαμε να υποστηρίξουμε το διάβημα το οποίο προτείνει ο εισηγητής. Εσείς ως πρόεδρος της Επιτροπής, πρόεδρε, να δείξουμε ότι στο κοινό, στην κοινή γνώμη, ότι ανεξάρτητα πολιτικού φάσματος όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποστέλει ένα χειρό μήνυμα σε ό,τι αφορά την προσχώρηση την πρόσβαση συγγνώμη, στα έγγραφα αυτά και την μη πολιτικοποίηση, αν θέλετε, της προσχώρησης στο Σέγγεν. Ευχαριστώ, κύριε Άλβαρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν συντομία, γιατί συμφωνώ ουσιαστικά με τον κύριο Κοέλιο. Απλά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο παράλληλα να τονίσουμε ότι Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει νομικό ενδεχομένω πλαίσιο μεταξύ του τι απαιτείται για προσχώρηση στη ζώνη Σέγγεν και άλλων ε, τομέων νομικής και μη συνεργασίας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη σύνδεση που υπάρχει. Και για να μην παρανοηθώ, θέλω να προσχωρήσει η Ρουμανία και η Βουλγαρία στη ζώνη Σέγγεν. Μην, μην πάρετε το τηλέφωνο κατευθείαν τον κύριο Πούτιν. Αυτό δεν χωράει εμφιβολία, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για δύο χώρες οι οποίες ε, στο δίκτυο διαφθοράς βρίσκονται πιο χαμηλά και από την Κούβα. Η μοναδική άλλη χώρα είναι η Ελλάδα. Άρα θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη ασκούν πίεση στις δύο χώρες αυτές να καταπολεμήσουν τη διαφθορά και είμαι βέβαιος ότι κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ των δύο θεμάτων. Καταλαβαίνω λοιπόν και εκείνους που ενδεχομένω να αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα στην παρούσα φάση. Και για να μην παραπονε... να παρανοηθώ, να πω ότι υποστηρίζω την προσχώρηση των δύο χωρών αυτών στη ζώνη του Σέγγεν, αλλά παράλληλα θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να μην ξεχνάμε που βρίσκονται ω προ τον δείκτη διαφθορά. Μάλιστα, Ο λέει ο πρόεδρο. Τώρα νομίζω ότι είναι η σειρά του Συμβουλίου να μιλήσει. Α, συγγνώμη κύριε Λάτφορντ, θέλετε κι εσεί το λόγο. Ναι, νόμιζα ότι με είχατε βάλει στο κατάλογο των ομιλητών. Φυσικά συμφωνώ με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα και να ευχαριστήσω τον Κάρλος και για τη μνήμη του, γιατί θυμάται τις προηγούμενες εμπειρίες και αυτό βοηθάει την Επιτροπή μας. Είναι χρήσιμο να ξέρουμε τι είχε συμβεί στο παρελθόν πριν από κάποια χρόνια. Και είναι λίγο εντυπωσιακό ότι έχουμε πάει προς τα πίσω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε λοιπόν όλες αυτές τις παρόμοιες εμπειρίες ε, διαφόρων προβλημάτων που είχαμε στο παρελθόν με το Συμβούλιο, είτε πρόκειται για πρόσβαση σε έγγραφα και αυτό δεν αφορά μόνο την Επιτροπή μας αλλά και το σύνολο του Κοινοβουλίου. Άρα νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα αναφέρουν όλα μαζί ο πρόεδρος Μπούζεκ, να αναφέρει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με το Συμβούλιο και για αυτά που είπε ο συνάδελφος Άλβαρο και νομίζω ότι το πάω και στην προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων. Νομικός, η αξιολόγηση αξιακή για τη ζώνη του Σέγγεν δεν καλύπτει θέματα που καλύπτει ε, ο μηχανισμός συνεργασίας που εφαρμόστηκε τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία το 2007. Και αυτό είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό ότι δεν υπάρχει τέτοια σύνδεση μεταξύ των δύο αυτών εγχειρημάτων. Το πρόβλημα όμω είναι ότι ο μηχανισμός αυτός δεν τροποποιήθηκε προκειμένου να αποτυπώνει αυτές τις ανησυχίες του 2007 και τώρα θα γίνεται ένας έλεγχος για τις νέες υποψήφιες χώρες που δεν είναι δυνατόν να επισέλθει σε αυτά τα θέματα. Και αυτό φυσικά καθιστά επιτακτική ανάγκη ο νέος μηχανισμός ελέγχου του Σέγγεν να καλύπτει θέματα όπως και τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ασφαλώς, αλλά και κακοδιαχείρισης και διαφθοράς. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες ανησυχίες σε μια ζώνη Σέγγεν όπου υπάρχει για παράδειγμα, παράδειγμα ανταλλαγή δεδομένων. Αλλά καταλήξαμε εδώ λόγω του μηχανισμού αξιολόγησης, πρώτης αξιολόγησης της ζώνης του Σέγγεν και ίσως δεν θα πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένος ο μηχανισμένος. Μάλιστα, ο κατάλογος ε, έκλεισε πριν από κάποια λεπτά, λέει ο Πρόεδρος, αλλά ξανανοίγει διαρκώ. Σας παρακαλώ, ε, συνεργαστείτε. Έγιναν πολλές προτάσεις, αλλά δεν υπάρχει κάποιο καινούργιο επιχείρημα για το βασικό ε, θέμα, για τη βασική πρόταση του κύριου Καέλιο, κύριε Παπα-Νικολάου, 30 δευτερόλεπτα και 30 δευτερόλεπτα για τον κύριο Μαρουνέσκου, αλλά νομίζω ότι καλό θα είναι να ακούσουμε και το Συμβούλιο. Κύριε Παπα-Νικολάου, ευχαριστώ, Πρόεδρε, ένα σύντομο σχόλιο. Και εγώ ασφαλώ υποστηρίζω αυτά που είπε ο κύριο Κοέλιο. Και όντω χρειάζονται συγκεκριμένα κριτήρια για να υπάρχει πρόσβαση στη ζώνη του Σέγγεν και θεωρούμε ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα τα καταφέρουν. Και φυσικά υπάρχει δείκτης για την διαφθορά. Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που είναι σε υψηλή θέση για την Ελλάδα, για τον δείκτη αυτό. Και νομίζω και άλλες χώρες ε, ε, είναι ψηλά σε αυτό το δείκτη. Μην αναφέρεστε λοιπόν μόνο συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Αυτό ως απάντηση στον κύριο Άλβαρο. Okay, and, and... Ο, ο Πρόεδρος. και δεν αναφερθήκατε και, δεν αναφερθήκατε και στην γλωσσική παραδρομή του κύριου Άλβαρο. Κύριε Μαρινέσκου τώρα εσείς. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες στατιστικές και βεβαίως ε, τα, αυτά που δείχνουν οι στατιστικές αληθεύουν. Τώρα το ερώτημα είναι πού πρέπει, σε ποια θέση πρέπει να βρίσκεται κανείς στατιστικές για να μπορεί να προσχωρήσει το Σέγγεν. Δεν θέλουμε να ε, διευρυνθεί η συζήτηση για να περιλάβει τώρα και τον ε, μηχανισμό συνεργασίας και Παλιθέψεως. Δεν υπάρχει άμεση διασύνδεση ανάμεσα στους δύο μηχανισμούς, ανάμεσα στο μηχανισμό αυτό δηλαδή και στον χώρο Σέγγεν. Για τον κύριο Άλβαρο μπορώ ευχαρίστως να του ε, διαβιβάσω πληροφορίες για τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην Ρουμανία, αλλά κύριε Άλβαρο θα πρέπει να αποφύγουμε να περιλάβουμε στην έκθεση τέτοιες, ε, τέτοια πράγματα ε, στην έκθεσή μας που λέει ότι άλλα κάνει η αστυνομία, άλλα κάνει η δικαιοσύνη και ό,τι καθεξής. Τώρα, ε, κύριε, κύριε Λούχαν, έχετε μόνο 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που δεν επιτρέπει την πρόσβαση στα έγγραφα αυτά το Συμβούλιο. Οι πολίτες απαιτούν να γνωρίζουν την αλήθεια. Πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν απολύτως πρόσβαση στα έγγραφα αυτά και να ζητήσουμε από τον πρόεδρο Μπούζεκ να ζητήσει με την σειρά του από το Συμβούλιο, εφόσον αυτό αρνείται, να αιτιολογήσει την άρνησή του. Καθώς επίσης να ζητήσει ο Πρόεδρος τον αποχαρακτηρισμό των ε, εν λόγω εγγράφων. Μέχρι τώρα δεν υπήρχαν τέτοια κριτήρια για τις χώρες οι οποίες ήθελαν να προσχωρήσουν στο ε, Σένγεν. Για ποιο λόγο άραγε να ισχύσουν αυτά μόνο για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ο πρόεδρος Αλβαρές βεβαίω θα το κάνουμε αυτό. Αλλά επιμένω ότι θα πρέπει να ακούσουμε τώρα την άποψη του Συμβουλίου και η εκπρόσωπός του είναι, είναι παρούσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος της Ουγγρικής Προεδρίας θα σας δώσω μια σύντομη επισκόπηση για το θέμα των εγγράφων. Τον Δεκέμβριο λάβαμε αίτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία υποβλήθηκε στο Κορεπέρ στις 20 Ιανουαρίου ελήφθη απόφαση, την οποία ανακοινώσαμε στο Συμβούλιο με επιστολή, πώς δηλαδή μπορούμε να εξασφαλίσουμε σε εσά πρόσβαση στα έγγραφα, σε έκτακτη διαδικασία πρόσβαση στα κτίρια μέσα του Συμβουλίου, στον Πρόεδρο, στους εισηγητές, συντονιστές. Δεν σας ικανοποίησε η πρότασή μας αυτή και γι' αυτό αναζητήσαμε νέες δυνατότητες, σας υποβάλαμε νέα προσφορά, την οποία επίσης δεν δεχθήκατε. Δεν τη δεχθήκατε την προσφορά, επικαλούμενη το γεγονός ότι θέλετε να υπάρξει μια οριζόντια λύση. Η Ουγγρική Προεδρία επεξεργάζεται τώρα τρίτη πρόταση την οποία στην επόμενη, στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας θα ε, θέσουμε υπόψη των δύο γενικών, αρμόδιων γενικών διευθύνσεων και έχουμε την πεποίθηση ότι έτσι θα λυθεί το θέμα. Καταβάλουμε διαρκώς προσπάθειες ώστε να μπορέσουμε να επιφέρουμε λύση. Ο πρόεδρος Άλβαρης, σας ευχαριστώ. Συγγνώμη, Αγγιλάρ. Ως πρόεδρος έχω διεξαγάγει και συνομιλίες με τον Ούγκρο μόνιμο εκπρόσωπο, μόνιμο αντιπρόσωπο και όλες οι προσπάθειες, σας διαβεβαιώ, έχουν γίνει από την Ουγγρική Προεδρία και τις εκτιμώ. Τις εκτιμούμε τις ε, προσπάθειες αυτές. Για να επιτευχθεί ο στόχος Δηλαδή να υπάρξει, να θεσπιστεί ένας τρόπος, ένας μηχανισμός ε, μιας αξιόπιστης συνεργασίας ανάμεσα στα δύο όργανα. Με τη λήψη μιας απόφασης πραγματικά αιτιολογημένης, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών να προχωρήσει τη σύνταξη νομοδότησης εν πλήρη γνώση των δεδομένων. Εκτιμούμε λοιπόν τις προσπάθειες που καταβάλει η Ουγγρική Προεδρία και θα τις εκτιμήσουμε βεβαίως απολύτως εφόσον επιτύχει το στόχο της και κάνει τη δουλειά της. Υπάρχει μια συμφωνία από ό,τι ε, μαθαίνουμε για την προθεσμία που θέλουμε να θέσουμε για την πρόσβαση στα έγγραφα με ορίζοντα τη Δευτέρα Μαΐου δηλαδή Εάν όμως εξακολουθήσει το Συμβούλιο να αρνείται την πρόσβαση στα έγγραφα, άκουσα και κάτι από τον κύριο Μαρινέσκου σχετικά με τον χρονικό ορίζοντα του Μαΐου. Ζήτησε λοιπόν να είναι νωρίτερα η προθεσμία αυτή, αλλά νομίζω ότι από ό,τι μαθαίνω δηλαδή υπάρχει συμφωνία μεταξύ σκιωδών εισηγητών και εισηγητού σχετικά με αυτό το νοδικό χάρτη που ε, μας εξήγησε ο κ. Κοέλιο. Άλλο πρόσθετο σχόλιο. Δέκα δευτερόλεπτα, λέει η κυρία Βέμπερ, σχετικά με αυτό που είπε η εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Προσέξτε, δεν είναι θέμα που θα λυθεί μεταξύ των γενικών γραμματέων των, ε, των ε, δύο οργάνων. Πρέπει οι πολιτικές ηγεσίε των οργάνων να αναλάβουν τις ευθύνες. Μα υπάρχει εδώ και πρόεδρος της Ένωσης. Δεν μπορούν να τα αποφασίζουν αυτά απλώς ανώτατη αξιωματούχη. βεβαίω, βεβαίω, έχετε δίκιο. Ο πρόεδρος Μπούσεκ. Γι' αυτό έχει κληθεί ο πρόεδρος Μπούσεκ να αναλάβει τα ενία τη υποθέσεω αυτή για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι αυτή τη φορά είναι αυτό το θέμα, αλλά εδώ διακυβεύονται πολύ περισσότερα. Ναι, συμφωνούμε λοιπόν. Θέλετε την τελευταία λέξη εσείς κύριε Κόλλιο. Ε, και θα είμαι σύντομο. Τρία σχόλια. Πρώτο. Τονίζω και υπογραμμίζω τα όσα είπαμε. Κι εγώ εκτιμώ τις προσπάθειες της Ουγγρικής προέδρια για την επίλυση του προβλήματος. Συναντήθηκα με τον πρέσβη, μίλησα στο τηλέφωνο με τον ε, υφυπουργό. Ξέρω ότι η Ουγγρική Προεδρία αναζητεί λύση και τους εύχομαι καλή επιτυχία. Γνωρίζουν ποια είναι η θέση της Ευρωβουλής και η συνεργασία των δύο οργάνων θα προσφέρει τη λύση. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμιά μακεβελική συνωμοσία ε, που ε, κάνουν πίσω από την πλάτη μας οι υπηρεσίες. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι η γραμματεία του Συμβουλίου δεν ενημέρωσε την Ουγγρική Προεδρία για τις συμφωνίες που είχαμε καταλήξει πριν από μία τετραετία. Άρχισαν τις διαπραγματεύσεις, αυτό μου έκανε εντύπωση, χωρίς να γνωρίζουν τι είχε προσφέρει το Συμβούλιο στο Κοινοβούλιο πριν από τέσσερα χρόνια. Και δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θα έπρεπε να τους είχαν εξηγήσει, να είχαν εξηγήσει στην Ουγγρική Προεδρία το επίπεδο εγγράφων στο οποίο είχαν προσφέρει πρόσβαση στο Κοινοβούλιο πριν από τέσσερα χρόνια. Τώρα, κάτι που είπε η κυρία Σοφή Ιντφέλτ. Συνήθως συμφωνώ μαζί της αλλά είπε τώρα ότι θα πρέπει να διατεθούν, να καταστούν δημόσια όλα τα έγγραφα. Εδώ δυστυχώς δεν θα συμφωνήσω. Από όσο γνωρίζω ορισμένε από τις εκθέσεις για την ασφάλεια και στα σύνορα αλλά και μέσα στο Σέγγεν, στο σύστημα Σέγγεν δηλαδή, δείχνουν ότι υπάρχει κάποια τροτότητα του συστήματος αυτό δεν μπορούμε να το καταστήσουμε δημόσιο κτήμα, διότι τότε παίζουμε το παιχνίδι των ανθρώπων που θα υποφεληθούν από την, τις αδυναμίες αυτές. Αυτό που ζητώ εγώ είναι αυτές οι ε, χαρακτηρισμένες εκθέσεις να τεθούν υπόψη των ευρωβουλευτών. Και τουλάχιστον στο επίπεδο που είχαμε πριν από τέσσερα χρόνια και όχι λιγότερα και βεβαίως κανονικά περισσότερα από τότε. Αν, αν δεν κατάλαβα καλά τι εννοούσε η Σοφή, τότε ζητώ συγγνώμη. Ε, ε, εάν δεν, ε, δεν ήταν αυτό που είπε η Σοφή και κατάλαβα λάθος, τότε, όπως είπα, ζητώ συγγνώμη. Τελευταίο σχόλιο για το όσα είπε ο κ. Μαρινέσκου. Εάν καταλήξουμε στις συνθήκες αν πληρούμε όλες τις συνθήκες για να παρουσιάσουμε την έκθεση πριν από τις 2 Μαΐου, τότε θα το πράξουμε. Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Μάρτιο ή Απρίλιο. Από τη στιγμή δηλαδή που θα πληρούνται οι συνθήκες. Δεν λέμε δηλαδή ότι θα υποβάλουμε την έκθεση μετά τις 2 Μαΐου. Είπαμε, εάν το Συμβούλιο δεν μας διαβιβάσει κανένα έγγραφο, δεν θα περιμένουμε πέραν από τις 2 Μαΐου γιατί πρέπει να βάλουμε κάποια προθεσμία μετά από την οποία δεν θα περιμένουμε άλλο. Αυτή ήταν η πρότασή μου και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Διευκρίνηση Ιντφέλτ. Ναι, όχι βεβαίω όλε ή λεπτομέρειε να καταστούν δημόσιο κτήμα, αλλά το κοινό έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιε είναι οι γενικέ γραμμέ, τα γενικά πορίσματα των έρευνών. Ο πρόεδρο Λόπε Αγγιλάρ. Νομίζω ότι η εκπρόσωπος του Συμβουλίου έχει, έχει σημειώσει τα διάφορα σχόλια και κυρίως την τελευταία δήλωση του κυρίου Κουέλιο. Και ας προχωρήσουμε τώρα στο υπαριθμόν 8. Επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφορικής. την απόρριψη του, την, ανάκληση της ε, Απόφαση πλαισίου του Συμβουλίου. Έχουμε εδώ τη συνάδελφο Μόνικα Χόλμαγερ. Αυτό το σημείο αφορά την προτινόμενη οδηγία για επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφορικής και την ανάκληση της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου για το θέμα. Το προτινόμενο κείμενο αναφέρεται σε ποινική νομοθεσία επί τη βάση του άρθρου 83 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κομισιόν τώρα λοιπόν θα μας κάνει μια πρώτη, ανταλλαγή, πρώτη παρουσίαση μάλλον και θα ακολουθήσει η συζήτηση αφού θα ακούσουμε την ησυχήτρια Χολμάιερ. Έχετε το λόγο κυρία Χολμάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα εδώ, και άμα καταφέρω, Κοιτάξτε, με κάποια θέματα μας απασχολούν ε, όταν άπτονται των δικών μας λογαριασμών, γιατί κοιτάμε θέματα επιθέσεων σε σελίδες του ίντερνετ και σε διάφορα τέτοια θέματα μετά την συζήτηση για το Wikileaks, όταν τα πιστοτικά ιδρύματα, οι τράπεζες ε, πλήχθηκαν, τα συζητήσαμε όλα αυτά. Ήταν μαζικές οι επιθέσεις κατά μεγάλων ε, επιχειρήσεων. Τότε έγιναν σαφείς οι επιθέσεις αυτές, οι απειλές αυτές. Η Γερμανία, η χώρα μου, Ε, κάθε μήνα έχει ένα εκατομμύριο δούρους ύπους που επιτίθενται σε κυβερνητικά συστήματα. Τα συστήματα αυτά ε, λειτουργούν μια χαρά, αλλά μιλάμε για ε, ζημιά 20 εκατομμυρίων ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Ένα σύστημα ασφάλειας κοστίζει σήμερα έσου και 250 ευρώ και καλωσορίζω λοιπόν ιδιαίτερα το γεγονό ότι υποβάλλει τέτοια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί με την ε, οδηγία αυτή θα έχουμε δυνατότητε ε, βελτίωση τη ε, άμυνά μα κατά των κυβερνοεπιθέσεων και κυρίω να κάνουμε και ευρωπαϊκά συντονισμένε δράσει. Εκ παραλλήλου, θα ήθελα να σα επιστήσω την προσοχή στο εξή. Η οδηγία αυτή δεν μπορεί παρά να είναι μια αρχή, μια κίνηση. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο ευρωπαϊκό πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε και να προβλέψουμε και μελλοντικά προβλήματα ενδεχομένω. Ένα παράδειγμα για κάποιε αδυναμίε. Ε, το cloud computing, όπως ονομάζεται στα αγγλικά, αλλά και κυβερνοεπιθέσεις κατά κρατικών συστημάτων, δημοσίων συστημάτων, μάλλον όχι μόνο κατά κρατών, αλλά και από κράτη, όπως για από την Κίνα, από τη Ρωσία και το καθεξής όπως έχει γίνει αντιληπτό. Και επίσης ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα του τι κάνουμε με τις επιχειρήσεις εκτός, είπα. Θα ήθελα να ακούσω και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα και κάποια σημεία τα οποία θα ήθελα να τα συζητήσω, κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε πριν από λίγο ότι ως τώρα αποτελούσε τη νομική μας βάση του άρθρου 80, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να, συζητάσουμε και, να συζητήσουμε και την πιθανότητα να κοιτάξουμε και το άρθρο για την αστυνομική συνεργασία για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού και χαίρομαι που θα συναντηθούμε, μάλλον ανυπομονώ να συναντηθούμε και με τους σκιώδες εισηγητές για να συζητήσουμε τις καλύτερες λύσεις για το θέμα αυτό και ανυπομονώ να ακούσουμε και τι έχει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, να ακούσουμε τι έχει να μας πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μας μιλήσει ο κύριος Γιάκοπ Μοντίνσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Είναι μεγάλη ικανοποίηση και χαρά για μας να παρουσιάζουμε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ την πρόταση της Επιτροπής για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφορικής. Είναι ένα από τα πρώτα βήματα της Κομισιόν για να ε, καλύψει τη νέα πραγματικότητα που δημιουργήθηκε μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας, άρθρο 83, παράγραφος 1. Είναι η πρώτη ουσιαστική πρόταση ποινικού δικαίου που προτείνει η Κομισιόν και όπως σωστά είπε η συγχύτρια, είναι ένα θέμα για το οποίο ακούμε καθημερινά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ίντερνετ αναμφίβολα αποτελεί πλέον ένα, μια σημαντική υποδομή της καθημερινής μας ζωής επί της οποίας βασιζόμαστε όλο ένα και περισσότερο. Εξαρτώμεθα από το ίντερνετ ε, στη δουλειά, ε, ως επιχειρήσεις, ως υπάλληλοι, αλλά και στην ιδιωτική μας ζωή εξαρτώμαστε, στην οικογενειακή μας ζωή επίσης. <coughs> Έχουμε δει ότι περιπτώσεις κυβερνοεγκλημάτων και κυβερνοεπιθέσεων είναι ένα άνευ συνόρων φαινόμενο και μάλιστα επεκτείνεται ζημιώνοντας τόσο την οικονομία όσο και με μονομένους πολίτες. αυτό, γι' αυτό χρειάζεται κοινή δράση από τα κράτη-μέλη σε επίπεδο της Ένωσης και μάλιστα είδαμε πως το θέμα του κυβερνοεγκλήματος έχει προχωρήσει σε διάφορα έγγραφα πολιτικής, στο πρόγραμμα Στοκχόλμης βεβαίως, αλλά τώρα έχει αναγνωριστεί ως και ένας από τους βασικούς στόχους προτεραιότητας στην εσωτερική, ε, στο εσωτερικό ανακοινοθέν που υιοθετήθηκε από την Κομισιόν τον περασμένο Νοέμβριο ε, ανακοινοθέν περί ασφάλειας. μεγάλο, ε, η για να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα ήταν ε, η επίθεση κατά της Εστονίας το 2007 και ε, κατά της Λιθουανίας το 2008. Το 2009 είχαμε ένα άλλο παράδειγμα που απέδειξε ότι τα πληροφορικά συστήματα κυβερνήσεων είχαν δεχτεί επιθέσεις σε 123 χώρες συμπεριλαμβανομένων και πρεσβειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελευταίους μήνες ακούσαμε για ένα νέο περίπλοκο ιό, το Stuxnet, το οποίο στόχευε σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η Europol πρόσφατα εξέδωσε την πρώτη αξιολόγηση απειλής όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα και το ίντερνετ που επιβεβαίωσε ότι οι εγκληματίες συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο ρομαντικών χάικερ, αν υπάρχει τέτοια κατηγορία, αλλά πάντως σοβαρές οργανωμένες εγκληματικές ομάδες χρησιμοποιούν το ίντερνετ. και το BOCnet είναι δίκτυα υπολογιστών που μπορεί κανείς να χειριστεί από, απόσταση για να ε, συντονίσει μια μεγάλη ε, επίθεση ταυτόχρονα. Και συχνά χρησιμοποιεί υπολογιστέ που αποτελούν μέρος αυτού του BOCnet όπως λέγεται, αλλά χωρίς να το γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες τους βασιζόμαστε στην ε, απόφαση πλαίσιο του 2005 και ακολουθούμε την ε, απόφαση, την εφαρμοστική για την απόφαση του 2008 που τόνιζε το γεγονός ότι ε, ένα νέο φαινόμενο είναι τα αυξανόμενα περιστατικά μεγάλη κλίμακας ταυτόχρονων επιθέσεων κατά πληροφορικών συστημάτων και η εγκληματική χρήση των BOCNET. Εμείς μέσω αυτής της οδηγίας θελήσαμε να στοχεύσουμε πολύ συγκεκριμένα, αλλά και να είμαστε και μετριοπαθεί για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα τέτοιο πλαίσιο για να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε τα κυβερνοεγκλήματα θα χρειαστεί μια μεγάλη διεθνής προσπάθεια, τουλάχιστον ευρωπαϊκού επίπεδου, Το κατάλληλο φόρουμ είναι η πεποίθησή μας ότι θα ήταν ε, η διάσκεψη των, ε, ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα και βασικός μας στόχος είναι να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες κλίμακες επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφορικής. Και σε αυτό βασιζόμαστε τώρα για να σας μιλήσω για τις βασικές διαφορές ανάμεσα στο απόφαση πλαίσιο και στην προτινόμενη οδηγία, να σας τονίσω κάποια σημεία. Στο άρθρο 6 εισάγεται ως ποινικό αδίκημα η παράνομη ε, ε, σύλληψη στοιχείων, ε, συλλογή στοιχείων, αυτό συνάδει με τη σχετική σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και στόχο έχει το άρθρο αυτό να προστατεύσει την την, τα ιδιωτικά δεδομένα την ε, ιδιωτική σφαίρα αλλά και την ε, διάθεση των ε, συστημάτων πληροφορικής και δεδομένων. Στο άρθρο 7 ποινικοποιείται η χρήση εργαλείων όπως το BOGNET, όπως το BOGNET που είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την διάπραξη του αδικήματος. Ποινικοποιούμε όχι μόνο τη χρήση αυτών, αλλά και την κατοχή, την πώληση ή την διάθεση, ώστε να αντικατοπτριστεί αυτό το γενικό παγκόσμιο φαινόμενο ειδικευμένων εγκληματιών που δεν ε, κάνουν οι ίδιοι τις επιθέσεις, αλλά ειδικεύονται στην παραγωγή τέτοιου είδους software και το πουλούν ή και το νοικιάζουν. Νοικιάζουν αυτές τις δυνατότητες σε άλλες εγκληματικές ομάδες. Στο άρθρο 9, η πρότασή μας αυξάνει το επίπεδο των ε, ποινικών κυρώσεων, ποινών. Ε, πιστεύουμε ότι αυτό δικατοπτρίζει το μέγεθος των κυβερνοκλημάτων, αλλά για μας είναι και ένα πολιτικό μήνυμα που προσδίδουμε ώστε να τονιστεί η σημασία της δίωξης αυτών των εγκλημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η minimum και η maximum ποινή είναι η φυλάκιση για ένα έως τρία χρόνια. Στο άρθρο 10 συμπεριλαμβάνουμε δύο δύο επιβαρυντικές περιστάσεις. Η πρώτη αφορά τη διάπραξη άλλων αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 6 μέσω της χρήσης του BOCNET. Και τα BOCNET που είναι μεγάλης κλίμακας. Δηλαδή προκαλούν σημαντική ζημιά ή ε, πλήττουν μεγάλο αριθμό υπολογιστών. Δεύτερη επιβαρυντική περίσταση είναι η κατάσταση όπου ο, οι ε, κλιματίες χρησιμοποιούν την ταυτότητα κάποιου άλλου για να κάνουν την επίθεση και μπορεί να προκαλέσουν σημαντική ζημιά στο συγκεκριμένο άτομο, δηλαδή το οποίο ε, χρησιμοποιούν την ταυτότητα. αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως κλοπή ταυτότητας. Αλλά λάβαμε συνείδητα την απόφαση να μην νομοθετήσουμε όπως στα υπόλοιπα ζητήματα ε, για την κλοπή ταυτότητας, αλλά για το συγκεκριμένο μόνο θέμα όπου η κλοπή ταυτότητας σχετίζεται με το κυβερνό έγκλημα. Άρθρο 14. Ε, είναι αυτό που εν μέρει απαντάει και στην παρατήρηση της εισηγήτριας. αφορά την ε, πρόθεση της συνεργασίας ανάμεσα στα κρατημέλη μέσω της επιβολής της υποχρέωσης να παρέχουν επίγοντος απάντηση μέχρι, μέσα σε 8 ώρες όταν δηλαδή υποβάλλεται έτοιμα βοήθειας. Έχουμε διαπιστώσει ότι τα σημεία επαφής ε, που λειτουργούν 24 ώρες το 24 ώρο δεν λειτουργούν τόσο αποτελεσματικά όσο θα το επιθυμούσαμε και πρέπει να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Και τέλος, το άρθρο 15 προβλέπεται υποχρέωση των κρατών μελών που στόχο έχει να δημιουργήσει μια κατάσταση όπου θα έχουμε συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για το κυβερνοέγκλημα σε ολόκληρη την Ένωση. Αναμφίβολα, μια από τις αδυναμίες της ε, μελέτης αξιολόγησης που έκανε η Κομισιόν ήταν το γεγονός ότι έπρεπε σε πολύ μεγάλο βαθμό να βασιστούμε σε στοιχεία από τη ΣΥΠΑ. Γιατί τα στοιχεία για την κατάσταση του κυβερνοεγκλήματος στην Ευρώπη είναι λιγοστά. Είναι ένα σημαντικό βήμα λοιπόν αυτό και άσχετα από την νομοθεσία που ισχύει τώρα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για να έχουμε ένα κοινό σύνολο δικτών ε, για να ξεκινήσουμε τη συλλογή στοιχείων. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτής της οδηγίας. Προσβλέπουμε σε επικοδομητική συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η σχετική συζήτηση στο Συμβούλιο έχει ξεκινήσει. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα, αλλά αναμφίβολα αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όπου από τη μια πλευρά τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν την ανάγκη εξυγχρονισμού των ισιών των μέσων, αλλά ταυτόχρονα ισχύουν συνήθεις ανησυχίες που προκύπτουν όταν μιλάμε ουσιαστικά για ποινικό δίκαιο με τα κράτη-μέλη, το επίπεδο των ποινών ας πούμε ή την ακαιρεότητα των νομικών ορισμών. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε πως το Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει τα νέα στοιχεία που έχουμε εισάγει και που, εν πάση περιπτώσει, αποτελούν μέρος των εντατικών συζητήσεων που γίνονται με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπορατίνσκι για αυτή την εισήγηση. Έχουμε κάποιους ε, βουλευτές που θέλουν να σχολιάσουν. Ο κύριος Άλβαρο είναι πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια δεκαετία μετά από τότε που είχε καταθέσει σχετική πρόταση το Συμβούλιο ε, έρχεται με δικές της προτάσεις. Ελπίζω να υπάρξει επικοδομητικός διάλογος. Παρακολουθώ το θέμα εκ μέρους της ομάδας μου και θα ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τον διάλογο αυτό. Α σκεφτούμε αν είναι η σωστή προσέγγιση το να ενταχθούν κάποιες παράγραφοι, κάποιες διατάξεις ποινικού δικαίου δεν ενδιαφέρουν πολλούς από τους χειριστές των Bognet που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε άλλες χώρες μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βοηθεί, τι θα βοηθήσει δηλαδή ε, το ποινικό δίκαιο εάν κάποιος έχει καταφέρει να παραλύσει ολόκληρη τη χώρα είτε, ούτε εάν αυξηθούν οι ποινές από ένα σε δύο ε, χρόνια για παράδειγμα στην Ισλανδία το 2007 είχαν παραλύσει 20.000 ε, ηλεκτρονικοί υπολογιστές τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα αυτοί που ενδιαφέρονται. Δεν τους ενδιαφέρει τώρα αν θα απειλούνται με φυλάκιση ενός ή δύο ετών. Ευχαρίστως λοιπόν να συζητήσουμε τα περί ποινικού δικαίου. Εγώ είμαι υπέρ ενός ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου, αλλά στην περίπτωση αυτή πραγματικά δεν μας προσφέρει τίποτα. Το άλλο πρόβλημα που βλέπω είναι σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των δικτύων πληροφορικής δεν πρέπει να τα βλέπουμε μονάχα αν υπάρχουν ε, το Wikileaks ε, που ε, για να υποστήριξουν το Wikileaks έριξαν κάποιες επιχειρήσεις που υποστήριξαν την Αμερικανική κυβέρνηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν σαφώς, σαφείς επιτιθέμενοι και σαφείς, σαφώς θύματα. Καμιά φορά τα παρακινούν και οι ίδιες οι κυβερνήσεις. Υπάρχουν λοιπόν hackers οργανωμένο έγκλημα, αλλά και κράτη ή δημόσιες αρχές, οι οποίες συμμετέχουν καμιά φορά σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι πώς θα εργαστούμε προληπτικά. Ωραία είναι να φροντίσουμε για ασφάλεια κτλ, Επιστευτικότητα των δεδομένων, όλα αυτά είναι σωστά. Αλλά πώς θα φροντίσουμε να υπάρχει προστασία από πριν. Το Stuxnet που αναφέρθηκε προηγουμένως, ο ιός που αναφέρθηκε προηγουμένως. οι αναλυτές αυτού του ιού καταλήγουν στην ε, πεποίθηση ότι 5 ή 6 άνθρωποι κάθισαν και δούλεψαν τουλάχιστον 5-6 μήνες και με πάρα πολλά λεφτά και φτιάξανε ένα ιό, ο οποίος μάλιστα μπήκε και ε, κάποιος δηλαδή αναγκαστικά πήγε σε μια εγκατάσταση πυρηνική των Ιρανών και την έβαλε σε ένα κομπιούτερ. Δεν ήταν κάτι το οποίο πέρασε μέσα από τα σύρματα. Τώρα, εκεί βλέπω πρόβλημα ασφάλειας. Και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε στην ε, Ευρώπη. Έχουμε ε, οργανισμό για ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων. Επίσης υπάρχει ο οργανισμός του ΝΑΤΟ που είχαν βοηθήσει για παράδειγμα στην περίπτωση της Ιρλανδίας που ανέφερα προηγουμένως. Η πεμπτουσία είναι η ασφάλεια των ε, πληροφοριακών συστημάτων είναι, πρέπει να είναι και φυσική και ε, τεχνολογική, όχι μόνο απέναντι σε ε, κακοποιούς, σε εγκληματίες, αλλά για παράδειγμα και σε αρχές άλλων χωρών. Υπάρχει συνεργασία. Προετών είχε γίνει μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής σχετικά με τη διαλειτουργικότητα. Εφόσον αυτό θα έχει επιληθεί το πρόβλημα, τότε θα μπορούμε να συνεργαστούμε. Για το λόγο αυτό, νομίζω ότι πρέπει λιγότερο να ε, προσπαθήσουμε να ε, στηρίξουμε την καταστολή, δηλαδή προς το, από το τέλος της διαδικασίας και περισσότερο την πρόληψη, που αυτή είναι το α και το ω για να αποφύγουμε τις δυσχέρειες αυτές δεν υπάρχει πλέον χρόνος να συζητούμε εάν θα υποστεί επίθεση η Ευρώπη, αλλά πότε και καμία χώρα δεν μπορεί να ισχυριστεί, η χώρα μέλος δεν μπορεί να ισχυριστεί στα σοβαρά ότι για παράδειγμα τραπεζικός της τομέας, ο δημόσιος της τομέας είναι επαρκώς ε, ασφαλής. Ευχαριστώ κύριε Φως. Ευχαριστώ. Είναι σωστή η προσέγγιση που ασχολούμαι τώρα με το cybercrime και τα λοιπά και μάλιστα εντατικότερα σωστά. Θα ε, συμφωνήσω και με τους συναδέλφους μου που ήδη μίλησαν. Πρέπει να κινηθούμε προς δύο κατευθύνσεις. Αφενός βέβαια την ποινική διάσταση, αλλά κυρίως βέβαια την προστασία απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις και επομένως πρέπει να τονιστεί και να τονωθεί πολύ περισσότερο η διάσταση της πρόληψης. Επίσης, στον τομέα αυτό, γιατί βέβαια το διαδίκτυο είναι και ένα παγκόσμια ισχύω μέσο, να δημιουργηθούν δια, που τέτοιες δεν έχουμε ακόμα μες στο σύστημα αυτό. Μία μικρή παρατήρηση τώρα σχετικά με το εξή. Για το μέλλον μου φαίνεται σημαντικό ίσως όχι απαραίτητα για την νομική πτυχή του θέματος, αλλά να διευκρινιστούν λίγο οι ορισμοί μεταξύ cybercrime και cyber war. Γιατί αυτά τα λεγόμενα phishing ή mobbing μέσα στο ίντερνετ είναι άλλη κατηγορία αδικήματος από την επίθεση κατά συστημάτων υποδομών κρατών ή ε, τραπεζικών συστημάτων ή ε, δημοσίων αρχών κλπ. Από την άποψη λοιπόν αυτή θα πρέπει να δώσουμε κάποιους ξεκάθαρους ορισμούς, ιδίως για παράδειγμα και διότι το ΝΑΤΟ στο νέο του δόγμα μιλεί και για κυβερνοπόλεμο. Επιθέσεις δηλαδή, ε, ηλεκτρονικές επιθέσεις κατά τραπεζικών συστημάτων για παράδειγμα. Αυτά νομίζω θα βοηθήσουν λίγο να διευκρινιστεί η εικόνα. Μιλντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει την προσπάθεια, διότι πρόκειται για σημαντική απειλή και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Εγώ είμαι αισιόδοξο αν αγοράσετε σήμερα ένα λάπτοπ θα δείτε ότι σε ένα χρόνο θα είναι απειρχαιωμένο, διότι οι εξελίξεις προχωρούν τόσο γρήγορα, μπορεί κανείς να τα προλάβει τα πράγματα αυτά. Μπορεί να υπάρξει ένας οργανισμός που θα αλλάζει τους κανόνες τόσο γρήγορα και τόσο συχνά. Χρειάζεται μια διαρκή συνεργασία, ε, ένας διαρκής μηχανισμός μάλλον, σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους τομείς. Μάλιστα, αρκετά σύντομος. Η κυρία Σιήτρια, η κυρία Χολμάιερ πάλι. Πρώτα, σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση του θέματος και των προθέσεών της. Δεύτερο, ευχαριστώ τον σκιώδη συγκητή μου για το γεγονό ότι έθεσε και το θέμα της ευρύτητας. Για παράδειγμα, μπορεί να βάλει κανείς μέσα και τα συστήματα αεροπορικών, συγκοινωνιών, ε, σιδηροδρομικών κλπ. Εξαρτώμεθα τόσο πολύ από την σωστή λειτουργία των δικτύων που πραγματικά δεν το συνειδητοποιούμε διαρκώς και παρόλα αυτά τα χρησιμοποιούμε καθημερινά διότι μπαίνουν σε κάθε τομέα της ζωής. Και για το θέμα αυτό που έφυξε ο Αλεξάνδρ Άλβαρο, για τα προληπτικά μέτρα δηλαδή, θα έλθω στο άρθρο 7 μέσα που χρησιμοποιούνται για το έγκλημα η εργαλεία η παραγωγή, πώληση, διάθεση στην αγορά, διάδοση και ούτω καθεξής τέτοιων οργάνων που χρησιμοποιούνται για την διάπραξη αδικημάτων. Αυτά περιλαμβάνονται λοιπόν εκεί στα σύγχρονα συστήματα. Υπάρχουν και συστήματα δοκιμασίας, τα οποία πρέπει πρώτα να λάβουν την έγκριση ότι επιτρέπεται να γίνει το τεστ. Θα χρειαστεί λοιπόν να ξανασκεφτούμε εάν η παράγραφος αυτή είναι σωστά διατυπωμένη. Διότι υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πρέπει να κάνουν τεστ για να διαπιστώνεται η ασφάλεια των συστημάτων μας, κινδυνεύουν να θεωρηθούν οι δράσεις τους αυτές αξιόπινες πράξεις. Αυτοί λοιπόν που ήδη εργάζονται δεν πρέπει να παρεμποδιστούν στην εργασία τους και ταυτόχρονα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον τα διάφορα ιδρύματα, Ινστιτούτα τα οποία ήδη υπάρχουν και λειτουργούν πολύ καλά για την ασφάλεια των ε, συστημάτων μας σε στενή συνεργασία με κρατικές αρχές και κρατικά ε, ιδρύματα μπορούν να δικτυωθούν καλύτερα διότι η συνολική αυτή προσπάθεια θα προσφέρει πολύ περισσότερα αποτελέσματα. Είμαστε στην αρχή της προσπάθειας βέβαια, το γνωρίζουμε και αυτό και η Κομισιόν το γνωρίζει και θα χρειαστούμε και τη συνδρομή πολλών εμπειρογνωμόνων από έξω. Σύντομα θα συγκαλέσω συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών και εμού για να κάνουμε και ένα σχεδιασμό και να ενισχύσουμε έτσι και τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία νομικού πλαισίου. Ευχαριστούμε κυρία Χολμάγερ. Νομίζω πως δεν έχουμε άλλα σχόλια. Να ακούσουμε ίσως κάποιες ε, παρατηρήσεις από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Παρακαλώ. Έχετε και πάλι τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ νομίζω πως ακούσαμε διάφορα κέρια σχόλια από τους ευρωβουλευτές σε σχέση με το θέμα του πώς μπορούμε να χειριστούμε το κυβερνοέγκλημα. Αναμφίβολα αυτό που σας παρουσίασα σήμερα είναι μια οδηγία ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Είναι δηλαδή ένα από τα διάφορα μέτρα πολιτικής που αναλαμβάνει η Κομισιόν. Δεν πρόκειται να είναι ένα κάτι το μαγικό που θα εξαφανίσει το πρόβλημα. Όχι, είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούμε να το ε, χειριστούμε. Γίνεται εντατική προληπτική εργασία. Πολύ αυτή εστιάζεται στην ε, αύξηση της γνώσης των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη για το πώς μπορούν να προστατευθούν από τον κίνδυνο επιθέσεων. Έχουμε επίσης ένα μεγάλο έργο που έχει ξεκινήσει ο Γενικός Διευθυντής Εξωτερικών Υποθέσεων με τη συνεργασία με την Europol για διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα. Πρόσφατα υπό την Ισπανική Προεδρία έχουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που προβλέπονται διάφορα μέτρα μεταξύ των οποίων και η δημιουργία ενός κέντρου Ευρωπαϊκού Κέντρου Κυβερνοεγκλήματος για το οποίο τώρα προετοιμάζουμε μια μελέτη σκοπιμότητας και στόχος το οποίο θα είναι να συντονίζει τις προσπάθειες των κρατών ε, μελών για την προστασία των βασικών υποδομών στον τομέα της ε, ε, τεχνολογίας της πληροφορικής. Όλα αυτά μπορούν κάπως να μας καθησυχάσουν ότι η απάντηση θα είναι κατάλληλη. Ωστόσο, θα τολμούσα να θυμίσω σε όλους μας ότι αυτό που θα συζητήσουμε στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας είναι βασικά Πενικές διατάξει. Ποινικό δίκαιο. Μια σημαντική διαφοροποίηση που πρέπει να γίνει είναι ότι χρησιμοποιούμε συνήθως το κυβερνόγκλημα με δύο έννοιες. Η μία και αυτό αντικατοπτρίζεται σε αυτή την οδηγία, είναι το στενό νόημα του κυβερνογκλήματο, είναι τα είδη εγκλημάτων που έχουν προκύψει ή που μπορεί να διαπραχθούν αποκλειστικά στο ίντερνετ. Ε, δεν υπήρχαν μπόκνετ. πριν να εμφανιστεί το ίντερνετ. Τώρα, για το phishing, το mobbing, αυτό είναι παραδοσιακά εγκλήματα τα οποία διευκολύνονται αυτή τη στιγμή από ε, το ίντερνετ. Το περίφημο ιός ε, της Νιγηρίας, το Nigeria Scam, ήταν, ε, λειτουργούσε εδώ και χρόνια, αλλά ήταν απλώς αποστολές γραμμάτων. Ε, τώρα όμως αυτά πολλοπλασιάζονται γιατί μπορούν να σταλούν με ένα, με ένα απλό email. Η οδηγία βέβαια ανταποκρίνεται και στον έλεγχο των συστημάτων ασφαλείας. Δηλαδή συγκεκριμένες ενέργειες είναι ε, αξιόπινες αν γίνονται μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Ας πούμε και οι εταιρείες ασφαλείας κάνουν ένα σώρο πράγματα για να ελέγξουν ε, την αντοχή των συστημάτων τους για παράδειγμα. Ελπίζω να σας βοήθησα με αυτές τις ευκρινήσεις. Σας ευχαριστούμε για την τελική αυτή παρουσίαση. Και νομίζω ότι αυτά αρκούν επί του παρόντος. Και έτσι λοιπόν προχωράμε στο 9. Το οποίο είναι και το τελευταίο σημείο επί της ουσίας το οποίο θα πραγματευτούμε σήμερα το απόγευμα. Μία ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους. Εδώ ο εισηγητής μας είναι ο συνάδελφος Βιν Φαντενκάμπ. Ο κύριο Φω, από ό,τι κατάλαβα, θα τον αντικαταστήσει. Να σα παρουσιάσω όμω το θέμα αυτό. Το θέμα αυτό αφορά την κατάρτιση μια νομοδότησης για μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίου σύμφωνα με μια πρωτοβουλία που έλαβε η Επιτροπή ΙΜΚΟ, η οποία και προετοιμάζει μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά που περιλαμβάνει 50 προτάσεις για να βελτιώσει τις εργασίες μας και τις ανταλλαγές. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το άρθρο 2 και για να, μπουν οι Ευρωπαίοι στο κέντρο της ενιαίας αγοράς. Θα μας μιλήσει λοιπόν ο κύριος Φως, ο οποίος εκπροσωπεί τον εισηγητή. Θα μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης και μετά θα έχουμε λίγα λεπτά για συζήτηση. Έχετε το λόγο κύριε Φως, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να σας ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του Wim ο οποίος δυστυχώς ε, είχε άλλες ε, σημαντικές ε, δεσμεύσεις. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ και γι' αυτό μου ζήτησε να παρουσιάσω το θέμα αυτό από πλευράς του. Έχετε μπροστά σας το σχέδιο γνωμοδότησης, πέντε στοιχεία περιλαμβάνονται και το θέμα είναι η αρμόδια επιτροπή για την ενιαία αγορά, μάλλον η Επιτροπή Ενιαίας Αγοράς και ιστορική και Καταναλωτή, να λάβει τις προτάσεις μας, προτού σχηματίσει την τελική τοποθέτησή της και εμείς από την πλευρά της Επιτροπής μας Χαιρετίζουμε φυσικά το γεγονός ότι υπάρχει η ανακοίνωση για την κοινή αγορά. Αυτό που μας δυσαρεστεί είναι ότι η εφαρμογή των προδιαγραφών αυτών δεν γίνεται σωστά από τα κρατη και γι' αυτό λοιπόν αφενός ζητάμε, απευθύνουμε έκκληση προς τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν τη διαδικασία της μεταφοράς και εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής και τα δεύτερον ε, ζητούμε να συμπεριληφθεί και να συμμετέχει καλύτερα ο Ευρωπαίος πολίτης στην πολυπλοκή αυτή διαδικασία για την ενιαία αγορά. Ζητούμε επίσης από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις σχετικές διατάξεις πιο γρήγορα και σε ό,τι αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες και κατά τέταρτον θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη αξιολόγησης της πρόοδου της εφαρμογής όλων των προδιαγραφών που έχουν προβλεφθεί για την ενιαία αγορά και στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη σαφήνεια και μεγαλύτερη ταχύτητα. Πέμπτο σημείο. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη σε ό,τι αφορά την εισρωή ε, μεταναστών υψηλής εξειδίκευσης, η οποία ασφαλώς είναι επωφελής για την ευρωπαϊκή οικονομία. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω βήματα σε ό,τι αφορά θέματα μετανάστευσης, πολιτικής ασύλου, σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες αυτές ομάδες. να βελτιωθεί η διαχείριση της μετανάστευσης ε, από το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ε, ληφθούν μέτρα για την πρόληψη της λαθρομετανάστευσης. Και θα παρακαλούσα λοιπόν τους συναδέλφους, ε, σε περίπτωση που έχουν παρατηρήσεις ή θέματα τα οποία θα ήθελα να συζητήσουμε, να μας τα πούν για να τα λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο, Ευχαριστώ, κύριε Φω. Και τώρα να μα μιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Μπερζέ. Θέλετε να πάρετε το λόγο εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Yes. Merci, merci, Monsieur le Président. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να υπενθυμίσω ορισμένα σχετικά με την ε, διαδικασία και τις προσδοκίες του κυρίου Μπαρνιέ πιο συγκεκριμένα. Έχει υποβάλει το σχέδιο πράξεως στις 27 Οκτωβρίου για μια ε, συζήτηση η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Την επόμενη εβδομάδα 8 Φεβρουαρίου στο κτίριο Σαρλεμάνι της Κομισιόν διεξάγεται σχετική διάσκεψη. Συνεργαζόμαστε στενά με την Επιτροπή σας Εσωτερικής Ιενίας Αγοράς Προσπαθούμε να είμαστε σε επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ εφόσον αυτέ επιθυμούν να γνωμοδοτήσουν. Για μας το πιο σημαντικό επί του παρόντο είναι να μπορέσουμε να διεξαγάγουμε διάλογο σχετικά με την προτεραιότητα που θα λάβουν τα διάφορα μέτρα ώστε να παρασκευάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τελικό κείμενο που ε, θα εγκρίνει το, ε, ε, στο σύνολό της, συλλογικός δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Άνοιξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπω μονάχα λίγους πλέον ε, ε, βουλευτές της Επιτροπής ΛΥΒΕ αλλά οι επιζώντες ας πούν κάτι <laughs> μετά από μια ε, σκληρή μέρα. Πρόκειται για την ενιαία αγορά αγαθών αλλά και υπηρεσιών. Πριν από λίγα χρόνια ήταν ο κύριος Μπόλκεστάιν που είχε υποβάλει πρόταση για να κάνει μια πιο δυναμική ε, αγορά των υπηρεσιών στην ενιαία αγορά. Διερωτώ με αν θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάτι παραπάνω στον τομέα αυτό, διότι η εντύπωσή μου είναι ότι αυτόν τον τομέα πρέπει να τον ενισχύσουμε περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες και να τον μελετήσουμε περισσότερο από τη σκοπιά αυτή. Ευχαριστώ κύριε Μιλντέρ. Άλλο κανεί δεν επιθυμεί να λάβει το λόγο. Κύριε Φως, εσείς μια τελευταία παρατήρηση. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μίλντερ για την πρότασή σας. Όντω, είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει να ε, θέσουμε με μεγαλύτερη έμφαση. Πρόκειται μοναχά εντό εισαγωγικών για γνωμοδότηση επί εκθέσεως που κάνει άλλη αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και από όσο μπορώ να δω εγώ η άλλη αυτή συναρμόδια, η αρμόδια της Ουσίας Επιτροπή ε, βλέπει το θέμα αυτό με τον τρόπο που βλέπετε εσείς, από τη σκοπιά που το βλέπετε εσείς. Σας ευχαριστώ κύριε Φως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει να προσθέσει τίποτε άλλο. Καλύτερα, καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας μένουν μόνο τα διάφορα. Κοιτάξτε πόσα πράγματα έχουμε τώρα. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για την Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου, το μεσημέρι, στις 12. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ για τις 7 Μαρτίου για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης της ενιαίας αγοράς. Μιλώ πάντοτε που συζητήσαμε σήμερα. Ο κύριος Φως, ναι, σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίες συνεδριάσεων κλπ. Θα ήθελα να έρθω στις 14 Δευτέρου και στις 17 Τρίτου ε, και να τις προτείνω αυτές τις ημέρες δηλαδή κατ' εντολή της ομάδας μου. Γνωρίζω βέβαια ποιες είναι οι δυσκολίες για την έγκριση του χρονοδιαγράμματος, αλλά έχουμε και εμείς όμως τις δικές μας ανηλυμένες υποχρεώσεις και τον σχεδιασμό μας ως ευρωβουλευτές, ώστε εκ των υστέρων είναι πάντα δύσκολο να μπορέσουμε να τα ρυθμίσουμε έτσι ώστε να μπορούμε να, να, μπορούμε να είμαστε παρόντες. Επίσης, θα ήθελα να δηλώσω το ότι δεν είμαστε σύμφωνοι να μεταφέρω τα πράγματα αυτά στο Στρασβούργο όλο και περισσότερο. Προτιμούμε να γίνονται στις Βρυξέλλες. Και αν ξαναγίνει πέμπτη θα δούμε παρόμοια, παρόμοιους αριθμούς παρόντων βουλευτών όπως τώρα που νομίζω ότι είμαστε τρεις όλοι και όλοι. Και δεν είναι σωστό να καταλήξει η διαδικασία αυτή σε χρονικά σημεία όπου δεν είναι πλέον δυνατόν να γίνει συζήτηση. Νομίζω ότι δεν, είναι, δεν ανταποκρίνεται στη σημασία του θέματος να διεξάγεται συζήτηση δηλαδή σε χρονικές περιόδους όπου οι περισσότεροι ήδη έχουν φύγει. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Και είμαι μάλιστα και ο πρώτος που, που ανησυχώ ε, λόγω της υπερεπιβαρημένης ατζέντα της ε, ε, Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών που είχε τρεις συνεδριάσεις αυτή την εβδομάδα και είμαστε η μοναδική επιτροπή που διεξάγουμε τακτικά, θα έλεγα, έκτακτες συνεδριάσεις και συνεδριάζουμε και στο Στρασβούργο. Έχουμε πρόβλημα με τον φόρτο εργασίας. Σημειώνουμε πάντως την ε, σύσταση που μας κάνατε για τις ημερομηνίες και το σημειώνω ότι τα λέτε αυτά εκπροσωπώντας τον κύριο Τικάμπ και το ε, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θα σας απαντήσουμε γραπτός, διότι φοβούμεθα ότι θα έχουμε πρόβλημα με το χρονοδιάγραμμα. Διότι πρέπει να συνδυάσουμε τη δική μας πορεία με αυτήν της ε, Επιτροπής ΙΜΚΟ που ψηφίζει στη τελική ψηφοφορία στις 7 Μαρτίου. Για να έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να ακουστεί η γνωμοδότησή μας, να είναι χρήσιμη λοιπόν, η μόνη λύση είναι 28 ε, Φεβρουαρίου. Θα σας απαντήσουμε γραπτός πάντως ε, σχετικά με τις προθεσμίες. Και πάλι λοιπόν θεωρώ ότι ήταν μια φορτωμένη εβδομάδα. Η επόμενη συνεδρίαση έχει ως εξής 14 Φεβρουαρίου. από 19 και 15 έως 21 βραδινές ώρες στο Στρασβούργο. Πάλι έκτακτη συνεδρίαση. Πάλι λοιπόν έκτακτη συνεδρίαση μέσα στην περίοδο συνόδου του Στρασβούργου. Μετά Φεβρουαρίου 28 από τις 3 μέχρι τις 4.30 αλλά τώρα λέει ο πρόεδρος μέχρι τις 6.30 ε, που όμως ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί στις 16 Μαρτίου στις 3 πάλι για 3.30 ώρες στις Βρυξέλλες και στις 17 Μαρτίου από τις 9 μέχρι τις 12.30 και από τις 3 μέχρι τις 6.30 πάλι στις Βρυξέλλες. Αυτά για την ώρα. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ευχαριστώ τους λιγοστούς επιζήσαντες, η κυρία Ζίπελ και ο κύριος Φως και καλό σας Σαββατοκύριακο.